κάποιες ανακοινώσεις, ε, θα τα διαβάσω στα τσεχικά. Ο Βίκτορ Σπάσκης μου μίλησε για τις ε, τελευταίες εξελίξεις και μου έχει στείλει ένα αίτημα για αναθεώρηση της απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου από τις 2 Σεπτεμβρίου του 2010 σχετικά με το καθεστώς ασυλίας του και αυτό το αίτημα θα το προωθήσουμε στην Επιτροπή Νομικών Υποθέσεων που είναι υπεύθυνη για τα θέματα αυτά. Η δεύτερη ανακοίνωση που ήθελα να σας κάνω ε, είναι ότι στις ε, 20 Ιουνίου συζητήθηκε η έκθεση Νάιτζερ Φαράζ από την Επιτροπή Νομικών Υποθέσεων και ο κύριος Νάιτζερ Φαράζ διαμετρήθηκε για, το θέμα, για την μεταχείριση του θέματος της ασυλίας του στην Ευρώπη. 11 μέλη ήταν υπέρ και 3 μέλη ήταν κατά. Δεν είναι παραδεκτό το αίτημα του κυρίου Φαράζ, διότι δεν τίθεται το θέμα ασυλίας του. Συνεχίζουμε λοιπόν αύριο, Τρίτη, 5 Ιουλίου, από τις 9 μέχρι τη 1 και από τις 3 μέχρι τις 8 και από τις 9 μέχρι τις 12 τα μεσάνυχτα. Η μερίσια διάταξη είναι στη διάθεσή σας και στην ιστοσελίδα μας και ολοκληρώσαμε την απόψινή συνεδρία. Σας εύχομαι καλό σας βράδυ και ευχαριστώ για την καλή σας συνεργασία. Και ευχαριστώ γενικά και τους διερμηνείς ο Πρόεδρος. Ευχαριστούμε.